Good evening. We'll start this meeting. First of all, I would like to say that Mr. Danjan, chairman of SEDE, could not be present today and he... Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ντανζάν, δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα και ζητά συγγνώμη. Υπάρχουν ορισμένες γλώσσες που δεν είναι διαθέσιμες σήμερα, δανέζικα, φιλανδικά, σουηδικά, Λετωνικά, σλοβενικά, μαλτέζικα, βουλγαρικά, τσεχικά, σλοβακικά και εσθονικά, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι η προτεραιότητα για διευμηνία έχουν οι γλώσσες των τακτικών μελών. Η αυριανή συνεδρίαση είναι βεβαρημένη ημερήσια διάταξη και θα ξεκινήσουμε ακριβώς στις 9. Αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις θα θεωρήσω την ημερήσια διάταξη δεκτή. Τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν και αυτά δεκτά. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τον αντιστράτηγο David Λίκη. Ο αντιστράτηγος είναι τακτικός επισκέπτης της Επιτροπής μας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νομοθετικής περίοδου και έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες εκ των έσω σχετικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τσάδ και στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Ο αντιστράτηγος πριν αναλάβει τη θέση αυτή ήταν υπεύθυνο για τη στρατιωτική δύναμη της Ένωσης στη Βοσνία ανάμεσα σε άλλες αποστολές που είχε αναλάβει. Μετά από τρία χρόνια θα παραδώσει τη διοίκησή του στρατιωτικού προσωπικού στον Φανχόχ από την Ολλανδία. Το στρατιωτικό προσωπικό, όπως γνωρίζετε, είναι η μοναδική στρατιωτική μόνιμη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την δυνατότητα να ενημερώνεται σε στρατιωτικό επίπεδο ο ύπατος εκπρόσωπος για τα εξωτερικά θέματα, έγκαιρη προειδοποίηση και αξιολόγηση κινδύνων. οι σημαντικές, δύο σημαντικές επιχειρήσεις ε, εξελίχθηκαν, η μία στο Τσάβ, κάτω από ένα πάρα πολύ εχθρικό κλίμα και η πρώτη ναυτική επιχείρηση, η Αταλάντα, κατά της πειρατείας στην περιοχή του Άντεν και στη Σωματική Ακτή. Κατά τη διάρκεια της διοίκησης του κυρίου Λίκη αναπτύχθηκε και η ιδέα του ευρωπαϊκού ε, στρατιωτικού σχηματισμού. Όπως ακριβώς είχαμε κάνει και με τον στρατηγό Τζέντε και θα πρέπει τώρα να ακούσουμε τις εντυπώσεις σας μετά από τρία χρόνια στη θέση αυτή. Θα θέλαμε επίσης ε, και να μας μιλήσετε για τη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σχέση σας με τη νέα προτινόμενη εξωτερική υπηρεσία. Θα θέλαμε επίσης να μας δώσετε τις απόψεις σας για τις καινοτομίες οι οποίες ε, γεννήθηκαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως η δομή μόνιμης συνεργασίας και το λεγόμενο ε, Ταμείο Startup. Θα θέλατε να μας μιλήσετε επίσης και για τις στρατιωτικές ικανότητες που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μελλοντικές επιχειρήσεις και για τους στρατιωτικούς μηχανισμούς, ε, σχηματισμούς που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Αντιστράτηγε, έχετε το λόγο. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά είμαι πάλι ανάμεσά σας. Αναφερθήκατε ότι ίσως είναι και η αποχαιρετιστήρια επίσκεψή μου γιατί στο τέλος του μηνός Μαΐου παραδίδω. Θα θυμίζω ότι σαν συνταξιούχος θα μπορούσα να σταθώ υποψήφιος βουλευτής και να έρθω εδώ με άλλη ιδιότητα. Απ' την άλλη βέβαια αυτή της τράπεζας. Πάντως σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Ελπίζω να καλύψω τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Θα ομαδοποιήσω τις παρατηρήσεις μου και δεν θα μιλήσω για πάνω από 20 με 30 λεπτά έτσι ώστε να μπορέσετε να θέσετε ερωτήσεις. Θα μιλήσω κυρίως για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν στρατιωτικός που υπηρετώ στο, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένιωσα πάντα ότι ο βασικός μου ρόλος είναι να δώσω τη δυνατότητα λειτουργικής επιχειρησιακής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου, θα έλεγα, υπηρεσίας, αυτό που έχει σημασία θεωρώ πάντα ότι είναι οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σημαντικό και θα αναφερθώ στα θέματα στα οποία πάντως εσείς αναφερθήκατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Θα μιλήσω καταρχάς για την επιχείρηση Αταλάντα. Δύο-τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις για την επιχείρηση Αταλάντα. Πρώτον, είναι η πρώτη θαλάσσια επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη, και μπορεί να σας εκπλήξει αυτό, είναι μια προσεκτική πολιτική στρατιωτική επιχείρηση και όχι μόνο στρατιωτική και αυτό δεν το έχει αναγνωρίσει ο περισσότερος κόσμος. Και τρίτον, είναι μια επιχείρηση η οποία αποδίδει μετρήσιμους καρπούς και είναι ιδιαίτερος χρήσιμη στην διεθνή κοινότητα διότι δίδει εγγυήσει και συνεισφέρει στην ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών ζωτικών για τις οικονομίες μας και το εμπόριό μας. Βασικός ρόλος αυτής της επιχείρησης, της στρατιωτικής επιχείρησης, της δύναμης ΝΑΒΟ, είναι να συνοδεύει ε, τα πλοία τα οποία μεταφέρουν Ε, τρόφιμα και υλικό ε, στην, ε, στις, στις ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρίσκονται στην Αφρική. Αυτή η προσπάθεια έχει στεφθεί από επιτυχία κατά 100% σε αυτή τη βασική αποστολή την οποία έχει η Αταλάντα. Έχουν υπάρξει 64 πλοία τα οποία έχουν συνοδευτεί και άλλα 32 διαφορετικής κατηγορίας χωρίς κανένα επεισόδιο σε ε, μια περιοχή ιδιαίτερως εχθρική. Αυτό σημαίνει ότι άνω των 300.000 τόνων τροφίμων έχουν παραδοθεί που έχει βοηθήσει στο να τρέφονται άνω των 6 εκατομμυρίων σωμαλών ημερησίως. Πρόκειται δηλαδή για μια βασική βοήθεια την οποία παρέχει το ναυτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν 20.000 πλοία τα οποία περνούν από τον κόλπο του Άντεν σε ετήσια βάση. Ήδη από τον Ιούλιο του 2009 μόνο δύο επιτυχείς επιθέσεις ολοκληρώθηκαν στον κόλπο του Άντεν και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποδοθεί μόνο στη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε όλες τις ναυτικές δυνάμεις που συνεισφέρουν στην ασφάλεια της περιοχής. Υπάρχουν επίσης άλλα 10.000 πλοία που χρησιμοποιούν άλλα τμήματα του Ινδικού ωκεανού, εκεί όπου καλύπτεται βέβαια από την Αταλάντα, και μόνο ένα πλοίο έχει, ε, θα έλεγα, ε, υποστεί πειρατεία. Και υπάρχει μια ιστοσελίδα ε, της Ευρωπαϊκής Ναυφός ε, για την θαλάσσια ασφάλεια ε, του κέρατος της Αφρικής που δίδει πληροφορίες ε, για την προστασία των πλοίων αυτών όχι μόνο βέβαια από τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις συμμαχικές θαλάσσιες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, των Ιαπώνων, των Ινδών και των Ρώσων. Πρόκειται λοιπόν για μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Αυτό το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι ότι μόνο ένα εμπορικό σκάφος έχει καταγραφεί ότι ε, έπεσε θύμα πειρατείας στην ιστοσελίδα. Όλα τα άλλα πλοία και ακόμα και αυτό το ένα, το οποίο έχει επαναλαμβάνω καταγραφεί, όλα αυτά τα πλοία λοιπόν, τα οποία έχουν υποστεί επιθέσεις, δεν ακολούθησαν τις βέλτιστες θαλάσσιες ναυτικές πρακτικές καταπολέμησης της πειρατείας. Οι πρακτικές αυτές είναι καταγεγραμμένες στην ιστοσελίδα NAFOR της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τους διεθνούς οργανισμούς ναυτιλίας, το IMO δηλαδή, σε συνεργασία με τις ε, εφοπλιστικές εταιρείες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έπρεπε λοιπόν να υπογραμμίσω ότι αν όλα τα πλοία της περιοχής ακολουθούσαν τις βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές και αν όλα τα πλοία ε, είχαν καταγραφεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαμε λιγότερα θύματα πειρατείας. Το δεύτερο μείζον σημείο είναι το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συντονισμού και διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις διεθνείς δυνάμεις που επιχειρούν στον Ινδικό ωκεανό. Εδώ νομίζω ότι εξηγείται αυτό και είναι η εξήγηση θα έλεγα ένα παράδειγμα της αρχής της πολυμερούς συνεργασίας σε πρακτική. Πάρα πολύ συχνά γίνεται μια συζήτηση για το αν αυτές οι θαλάσσιες ε, οι ε, μορφές προστασίας θα πρέπει να αναλαμβάνονται από το ΝΑΤΟ ή από ομάδες χωρών προθύμων να το κάνουν ή από, μόνο, από μόνη της την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά η συνεργασία αυτών των τριών επιπέδων έχει διευκολύνει κατά πολύ τα πράγματα και έχει επιτρέψει σε άλλες χώρες με θαλάσσιες στρατιωτικές δυνάμεις να συνεισφέρουν με τα δικά τους πολεμικά σκάφη στα πλαίσια της συντονιστικής ομπρέλας του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμμαχίας Ναυτικών Δυνάμεων. Έχει σημασία λοιπόν το ότι μόνο όταν το ευρωπαϊκό κομμάτι αυτής της θαλάσσιας δύναμης συγκεκριμένα προσκάλεσε τους Ιάπωνες, τους Κινέζους και τους Ρώσους και τους Ινδούς να πάρουν μέρος σε αυτή τη μορφή συνεργασίας. Μόνο λοιπόν όταν εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αποστήλαμε αυτή την πρόσκληση και όχι οι Βρυξέλλες αλλά οι διοικητές των ναυτικών δυνάμεων τότε αυτές οι χώρες ήλθαν και συμμετείχαν και ε, εφάρμοσαν το πρόγραμμα SHADE, το οποίο είναι το πρόγραμμα α, από κοινού συνειδητοποίησης ε, των κινδύνων. Είναι συλλογή πληροφοριών το πρόγραμμα αυτό, γίνεται αντικείμενο συντονισμού από τις ναυτικές δυνάμεις, επαναλαμβάνω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και η Κίνα επίσης αναλαμβάνει έναν σημαντικά καθοριστικό ρόλο. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα πολυμερούς συνεργασίας η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη και πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό. Το τρίτο σημείο, το έχω ήδη πει σύντομα στην εισαγωγή μου, είναι η συνολική ε, φύση της ε, επιχείρησης Αταλάντα. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια αυστηρά ναυτική επιχείρηση. Προφανώς εμπλέκει και αεροσκάφη όμως. Και τα αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αποστολή αυτή είναι πραγματικοί πολλαπλασιαστές δυνάμεως λόγω της δυνατότητας ελέγχου που έχουν και της ταχύτητας με την οποία καλύπτουν τεράστιες περιοχές. Αλλά υπάρχει και ο πολιτικός τομέας ο οποίος είναι εντυπωσιακό. Αν μπείτε στο στρατηγείο στο Northwood της Αγγλίας, όπως το κάνω συχνά, θα δείτε αυτό το οποίο περιμένετε. Δηλαδή ε, πάρα πολλούς αξιωματικούς του ναυτικού με πάρα πολλούς ε, ε, υπολογιστές, κάποιους αξιωματικούς του στρατού και της αεροπορίας, αλλά και πάρα πολλούς με πολιτικά. Όχι με κουστούμια, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι με στολές. Ναι, ναι. Με πολιτικά, πολιτικές στολές, λέει ε, ο κύριος Λίκη. Έχω συνηθίσει όταν πηγαίνω σε στρατητικές εγκαταστάσεις και βλέπω πολλούς κόσμους με πολιτικά, είναι συνήθως πολιτικοί και νομικοί σύμβουλοι. Και μου έκανε εντύπωση πως οι νομικοί σύμβουλοι δεκάδες ήταν εκεί με πολιτικά. Και φυσικά με διόρθωσαν. Και μου είπαν ότι αυτοί δεν ήταν Paul Ads και League ads ήταν της ε, ε, εφοπλιστικής κοινότητας, ε, της αλλιευτικής κοινότητας και συμμετείχαν στην, στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων στο Northwood. Δηλαδή συνδυασμός των ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων και των πολιτικών δυνάμεων που εμπλέκονται στην ιστορία αυτή. Σύντομα τώρα να αναφερθώ στα κράτη-μέλη τα οποία συνεισφέρουν στην ε, ε, επιχείρηση αυτή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη Γαλλία. Δεν ακούτε έναν Άγγλο αξιωματικό να επενεί τη Γαλλία τόσο συχνά. Αλλά η Γαλλία σε κάποια φάση είχε 14 πλοία σε αυτήν την επιχείρηση. Και είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω τις χώρες οι οποίες έχουν δώσει και περιπολικά αεροσκάφη Λουξεμβούργο, Ισπανία, Γαλλία, Σουηδία και Ισπανία. Γιατί τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας είναι οι πραγματικοί πολλαπλασιαστές της ναυτικής δύναμης καλύπτοντας τεράστιες περιοχές. Λίγα ακόμα λόγια για την Αταλάντα. Καταρχάς με τους πειρατές οι οποίοι είχαν συλληφθεί και κάποιες στατιστικές για το τι συμβαίνει μετά το τέλος των μουσώνων. Όταν δηλαδή ξαναρχίζει η πειρατική δραστηριότητα μετά το τέλος των μουσώνων, των τροπικών καταιγιδών. Ε, τις τελευταίες ε, τρεις-τέσσερις εβδομάδες μετά από το τέλος της εποχής των μουσώνων έχει υπάρξει ένας ειδικά υψηλός αριθμός πειρατικών ενεργειών οι οποίες ε, εμποδίστηκαν από την ναυτική δύναμη. Να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Και αυτό αφορά τα στοιχεία στα οποία εμπλέκονται τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι των υπολείπων δυνάμεων. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι έχουν ε, πέσει θύματα πειρατείας, επιτυχούς πειρατείας, τρία πλοία και άλλα τρία αφέθηκαν. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ισορροπία στην εφοπλιστική δραστηριότητα. Από την άλλη όμως 11 πειρατικές ενέργειες διεκόπησαν, παρεμποδίστηκαν 11. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Σομαλίας. Αυτό σημαίνει ότι πέντε πλοία μητέρες, πέντε πλοία δηλαδή από τα οποία εξαρτώνται μικρές, τα μικρά πλοία των πειρατών καταστράφηκαν. 67 πείρατες ε, συνελήφθησαν, 11 από αυτούς θα σταλούν στις Εχέλες και θα διωχθούν εκεί μετά από μια λογική συμφωνία την οποία συνήψαμε με την κυβέρνηση των Σεϊχελών για τη δίωξη των πειρατών. Από τους υπόλοιπους πειρατές οι οποίοι κρατούνται αυτή τη στιγμή 56 θα απελευθερωθούν ή έχουν ήδη απελευθερωθούν, απελευθερωθεί συγγνώμη, γιατί δεν είχαμε αρκετά ισχυρές αποδείξεις έτσι ώστε να τους παραπέμψουμε σε δικαστήριο και να δικαστούν. Συνεπώς νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με καλές επιδόσεις. Έχουμε επίσης και μια συμφωνία μεταφοράς στην Κένια, με την Κένια έτσι ώστε κάποιους από τους πειρατές να τους δικάσουμε στα πλαίσια της κενιατικής δικαιοδοσίας. 75 πειρατές έχουν αποσταλεί στην Κένια, από τους οποίους οι 8 καταδικάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και άλλοι 9 αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δικάσιμη διαδικασία. Λοιπόν, θα κλείσω με την Αταλάντα λέγοντας σύντομα κάποια λόγια σχετικά με την αποτελεσματικότητά της Υπάρχουν παρόλα αυτά εμπορικά πλοία που πέφτουν θύματα πειρατείας. Προφανώς ασκώ κριτική σε κάποια από τα πλοία αυτά γιατί δεν παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία είναι γνωστά της πάση. Από την άλλη όμως, εμείς που παρέχουμε τις θαλάσσιες και εναέριες δυνατότητες δεν μπορούμε να είμαστε φυσικά παρόντες παντού σε όλη αυτή την τεράστια ναυτική περιοχή. Αλλά το ποσοστό των επιτυχών πειρατικών ενεργειών έχει σταφέστατα μειωθεί σε σχέση με το 2008. Από το 2008 μέχρι το 2009 έχει υπάρξει μια συστηματική μείωση των πειρατικών ενεργειών, πόσο μάλλον που μόνο μία στις τέσσερις πειρατικές απόπειρες είναι πλέον επιτυχής. Βλέπουμε ε, να μειώνεται και ο αριθμός των πειρατών. Σας δίνω πάλι στατιστικές που αφορούν τη δική μας ναυτική δύναμη και όχι τις άλλες χώρες. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτης στην προσπάθεια αυτή, ακόμα και σε επίπεδο των πειρατών που έχουν συλληφθεί από τους Ρώσους, τους Ιάπωνες, τους Ινδούς, τον ΝΑΤΟ κτλ. Δεν θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες στρατιωτικές ναυτικές δυνάμεις. Αντίθετα, ο συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες ναυτικές δυνάμεις είναι εξαιρετικά καλός και είναι θέμα τύχης εν πωλής και όχι τόσο προγραμματισμού που σου δίνει τη δυνατότητα, που μας δίνει τη δυνατότητα να βρούμε τους πειρατές αυτούς. Είναι σαν να ψάχνει κανείς καρφίτσα στο άχυρο να βρει. Θα περάσω τώρα στην ε, επιχείρηση Άλτεα, την επιχείρηση σταθεροποίησης της Βοσνίας Ευζεγοβίνης. Η επιχείρηση αυτή συνεχίζεται με την εκτελεστική εντολή διατήρησης περιβάλλοντος ασφαλείας. Είναι επιτυχής μέχρι τώρα η επιχείρηση. Ο κίνδυνος ε, σύγκρουσης ή και ε, μικρότερο επίπεδου σύγκρουσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές κοινότητες αυτό δείχνει ότι υπάρχει και έλλειψη όρεξης για σύγκρουση από πλευράς των κοινοτήτων λόγω και ορισμένων εξελίσεων στον πολιτικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό τομέα. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια συνέπεια της ε, ε, διεθνούς κοινότητας η οποία συνεχίζει να εμπλέκεται στη Βοσνία Ευζεγοβίνη με τη στρατιωτική της δύναμη. Αυτή η στρατιωτική δύναμη αναγνωρίζεται με αλφαγιώτα και από τον είπα το εκπρόσωπο της Ένωσης στη Βοσνία, τον κύριο Ένσκο, ότι η στρατιωτική δύναμη λειτουργεί μετριαστικά, ηρεμιστικά θα έλεγα, σε ένα περιβάλλον πολιτικά και μάλιστα τώρα στην προεκλογική περίοδο ε, θα έλεγα σε ένα περιβάλλον πολιτικά σταθές και επικίνδυνο, Αναβράζουν πολύ θα έλεγαν θα πρέπει να διατηρηθεί η εκτελεστική αυτή έντολη μέχρι το τέλος τουλάχιστον της εκλογικής περίοδου ή μέχρι το τέλος του 2010 έτσι ώστε να συνεχίσουμε και μετά το 2010 αφού επανεξεταστούν οι συνθήκες. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει να αυξήσει αυτή την ε, προσπάθεια σταθεροποίησης και με μια εκπαιδευτική αποστολή η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την αντίστοιχη προσπάθεια την οποία επιτελεί το ΝΑΤΟ στο Σαράγεβο. Η εκπαιδευτική αυτή αποστολή την οποία θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπαιδεύει τους ε, Βόσνιους αξιωματικούς σε τακτικό επίπεδο, στο κατώτερο επίπεδο, σε επίπεδο υπαξιωματικών βασίζεται σε μια ανάλυση των αναγκών σε εκπαιδευτικό επίπεδο η οποία έχει γίνει ανάμεσα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις στρατιωτικές δυνάμεις της Βοσνίας Ευζεγοβίνης. Είναι μια ιδιαίτερα κακοφόρα προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν ανησυχίες βέβαια ότι δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη διαθέσιμα να διατηρήσουν τα επίπεδα των δυνάμεων που έχουν στη Βοσνία ερζεγοβινη αντίστοιχα με τα παρόντα και μετά την προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει χένον, αλλά νομίζω ότι είναι πολιτικό θέμα και δεν είναι ε, στρατιωτικό και δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Η τρίτη επιχείρηση, η οποία δεν είναι ακριβώς επιχείρηση αλλά είναι αποστολή θα έλεγα, και βρίσκεται στα τελικά στάδια προγραμματισμού και στο πρώτο στάδιο εφαρμογής, είναι η εκπαιδευτική αποστολή στη Σομαλία η οποία θα διεξαχθεί στην Ουγκάντα βέβαια. Στόχος αυτής της αποστολής είναι να συνεισφέρουμε στην κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας, οι οποίοι έρχονται από το Μογκαντήσου στην Ουγκάντα, έχουν ελεγχθεί από την ε, επιχείρηση Έμεσον, Έρχονται λοιπόν στην Ουγκάντα όπου οι δυνάμεις της Ουγκάντα έχουν ήδη εκπαιδεύσει σημαντικούς αριθμούς Σομαλών έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας και καταστολής ε, ε, και να υπό τον έλεγχο της μεταβατικής ομαλικής κυβέρνησης. Το πρόγραμμα αυτό θα ε, προβλέπεται να διαρκέσει ένα χρόνο ή περίπου ένα χρόνο. Πρέπει να συνεισφέρουμε στις επόμενες δύο σειρές Σομαλών χίλιοι κάθε φορά εκπαιδεύονται και η εκπαίδευση κρατάει έξι μήνες. Και μετά επιστρέφουν στο Μογκαντήσου και εκεί τίθενται υπό τη διοίκηση των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας. Στόχος λοιπόν είναι να εκπαιδεύσουμε δύο σειρέ, θα έλεγα αξιωματικών ή αξιωματούχων. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε ε, την κυβέρνηση της Ουγγάντα σε συγκεκριμένους τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι η ε, εκπαίδευση αξιωματικών και υπαξιωματικών έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα ε, στις σομαλικές αρχές να διαμορφώσουν μια ιεραρχία στο εσωτερικό τους, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα να εκπαιδεύσουμε ειδικέ δεξιότητες σε ορισμένους τομείς, όπως ε, οι επικοινωνίες, ή σύραξη σε εσωτερικό επίπεδο πόλεων, και διάφορε άλλε ειδικέ ενέργειε οι οποίε θα βοηθήσουν τι ομαλικέ δυνάμει καταστολής να γίνουν πιο αποτελεσματικέ. Η αποστολή αυτή νομίζω ότι θα ολοκληρώσει την προγραμματική της φάση και θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο και θα κηρυχθεί έναρξη λειτουργία της στο τέλος του μηνός Μαρτίου. Έχουμε ήδη μια μικρή ομάδα στην Ουγκάντα η οποία ε, κάνει ό,τι προπαρασκευαστικό χρειάζεται και ε, οικοδομή θα έλεγα τις τελευταίες υποδομές που είναι απαραίτητες για να ενισχύσουμε ε, τις ε, εγκαταστάσεις που έχουν ήδη δημιουργήσει στην Ουγκάντα η κυβέρνησή της. Οι αρχικές επιχειρησιακές ικανότητες αν θέλετε αυτής της επιχείρησης θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν στα μέσα Απριλίου και θα φτάσουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα στο τέλος του μηνός Απριλίου αρχές Μαΐου για να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση αυτών των σειρών Σομαλών. Αυτή η προσπάθεια συντονίζεται από την κυβέρνηση της Ουγκάντα, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι ενισχύουν και την παρουσία της επιχείρησης ένεσων στη Σομαλία. Θέλουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν την κυβέρνηση της Ουγκάντα δίδοντας επιπλέον εκπαιδευτές και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς που ανέφερα. Το μέγεθος αυτού του αποσπάσματος του εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ μικρό. Πρόκειται θα έλεγα για ένα μικρό κομμάτι όπου μια μικρή κοινοτική συνεισφορά παρόλα αυτά θα προσφέρει δυσανάλογα πολύ στην ασφάλεια της Σομαλίας η εκπαιδευτική αυτή θα, είναι, θα αποτελείται από μια δύναμη 140 ανδρών που δεν θα είναι όλοι μαζί όμως παρόντες. γιατί οι Σομαλοί όταν πηγαίνουν εκεί μένουν μερικές εβδομάδες ή και μήνες πριν είναι πλέον ικανοί να δεχθούν τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς αλλά οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί μάλλον θα εκπαιδεύονται εξ αρχής από τις ε, ευρωπαϊκές δυνάμεις. Επανέρχομαι λοιπόν σε εκπαιδευτικές ε, ε, παρεμβάσεις. Εδώ υπάρχει διοικητής Ισπανός συνταγματάρχης. Η Ισπανία είναι η ηγέτιδα δύναμης, η ηγέτιδα χώρα θα ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα με ποια επιχείρηση ασχολήθηκα τα τελευταία τρία χρόνια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν υπάρχει ένα κράτος μέλος το οποίο ε, θέλει να λειτουργεί σαν χώρα πλαίσιο ή σαν ηγέτης χώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο διευκολύνει τα μάλα τα, ε, την επίλυση ε, των προβλημάτων τα οποία αναδύονται και διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης και η Ισπανία παίζει ένα σαφέστατο ρόλο διευκολύνοντας τη συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια. Θα θίξω τώρα και κάποιους άλλους τομείς, τους οποίους εσείς αναφέρατε ότι θα πρέπει να, σχολιάσω και μετά θα περιμένω τις ερωτήσεις σας. Οι άλλοι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός μας στόχος είναι να διαμορφώσουμε και δυνατότητες αξιολόγησης και προειδοποίησης εγκαίρων, κινδύνων. Η ανταλλαγή πληροφοριών λειτουργεί σε σύγκριση 40 άτομα προσωπικό που ασχολούνται με αυτό και κάνουν αυτό το οποίο περιμένει κανείς, δηλαδή ελέγχουν σε επίπεδο πληροφοριών αυτά τα στοιχεία τα οποία παίρνουν. Το σύστημα λειτουργεί καλά αν σκεφτεί κανείς ότι οι πληροφορίες προέρχονται από 27 χώρες. Όπως ε, και με όλα τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα πάνε καλύτερα όταν γίνονται με συνολικό τρόπο. Όταν υπάρχει συνεργασία του πολιτικού τομέα και του στρατιωτικού τομέα. Και όταν συνδυάζονται οι αναλυτικές επιχειρησιακές δυνατότητες ε, των πολιτικών υπηρεσιών με τις στρατιωτικές δυνάμεις. Ε, πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Δεν διεκδικώ εγώ την επιτυχία αυτής της συνεργασίας. Υπάρχουν όμως ε, πολλοί άλλοι συνάδελφοι και υπάρχει ένας λιθούανό στρατηγός ο οποίος μέχρι τώρα ήταν υπεύθυνο για τη συνεργασία πολιτικού στρατιωτικού τομέα και γενικά η δυνατότητα η επιχειρησιακή συλλογής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Σε άλλους τομείς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας σε επίπεδο προσωπικού λειτουργεί σαν αναλυτές έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να ε, διαμορφώσουμε δυνατότητες τέτοιας προσπάθειας. Θα αναφερθώ σε κάποιους από τους τομείς τους οποίους υπάρχει μια προεργασία ήδη σήμερα. Αναζητούμε φυσικά πάντα να αναθεωρήσουμε και να επικαιροποιήσουμε κάποιες ε, έννοιες τις οποίες θεωρούμε σταθερές. Καταρχάς, η γρήγορη απάντηση, η γρήγορη αντίδραση, η ταχεία αντίδραση αν θέλετε. Ε, κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων προεδριών, της Ισπανικής και της Σουηδικής, έχει υπάρξει μια κάποια συζήτηση για τη χρησιμότητα των ευρωπαϊκών στρατιωτικών σχηματισμών. Έχουν γίνει συζητήσεις πάρα πολλέ και σε υπουργικό επίπεδο και θα ακούσατε και τις δηλώσεις της Σουαδικής Προεδρίας η οποία λέγει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση των σχηματισμών των στρατιωτικών. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, γιατί δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να υπάρξουν ορισμένες βελτιώσεις και υπάρχει αρκετή πρόοδος η οποία έχει συντελεστεί στα πλαίσια της ανάπτυξης της ε, έννοιας αυτών των σχηματισμών ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στα πλαίσια της βελτίωσης ή σμίκρησης, αν θέλετε, του χρόνου αντίδρασής τους. Παρενθετικά εδώ να πω ότι εκμεταλλευόμεθα τα μαθήματα που παίρνουμε και από την αιτή, από την εμπειρία της IT και τα εντάσσουμε ε, στις εικόνες χρησιμότητας που θα θέλαμε να δίνουν στο μέλλον οι σχηματισμοί αυτοί. Θαλάσσια ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Εξετάζουμε την έννοια αυτή της ασφάλειας στη θάλασσα και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας έχει ζητήσει από πέντε ναυάρχους και αντί ναυάρχους να προχωρήσουν στην διατύπωση μιας έκθεσης, στη σύνταξη μιας έκθεσης η οποία μόλις συμπληρώθηκε, ολοκληρώθηκε και βρίσκεται υπό εξέταση στη γραμματεία της ε, Υπηρεσίας Άμυνας. Πολλά γίνονται και στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας δηλαδή. Πολλά επίσης ε, έχουν προσφέρει εδώ η Ισπανική και η Σουηδική Προεδρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν οι δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για διάφορες επιχειρήσεις τύπου και πά. Υπάρχει ένα δίλημα για τους στρατιωτικούς όπως εγώ βέβαια, το οποίο παραμένει πάντα. Βλέπουμε ας πούμε τη, τη χρησιμότητα βελτίωσης της ικανότητας ναυτικής συνεργασίας, σαν παράδειγμα στη Μεσόγειο, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες μορφές πολυεθνικής συνεργασίας σε επίπεδο ναυτικής ενός συνεργασίας και ελέγχου. Όχι μόνο οργανώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα συλλογής πληροφοριών και το θέμα είναι σε ποιο βαθμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις και πά. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την τεχνολογία την διαθέσιμη και θα πρέπει να την μετατρέψουμε σε σύγχρονη τεχνολογία η οποία να χρησιμοποιείται εκτός Ευρώπης βέβαια και όχι εντός του ευρωπαϊκού εδάφους και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες και ικανότητες που έχουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε αν κάτι από αυτό θα ήταν χρήσιμο και στο εσωτερικό της Ένωσης. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι έχουμε συγκεκριμένες προκλήσεις αυτή τη στιγμή και πρέπει να καλύψουμε και τα προβλήματα πέρα από τον προγραμματισμό. η αρχιτεκτονική η ιεραρχική η αρχιτεκτονική ελέγχου αν θέλετε των επιχειρήσεων αυτών είναι θα έλεγα υπηροκεντρική δηλαδή αφορά περισσότερο χερσαίες επιχειρήσεις και η εμπειρία που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα είναι εμπειρία η οποία αφορά τις χερσαίες ακριβώς επιχειρήσεις. Έχουν σχεδιαστεί δηλαδή για να λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές. Και στον τομέα των θαλάσσιων επιχειρήσεων τα πράγματα ήταν πιο περίπλοκα. Πήραμε λοιπόν μαθήματα από τις αδυναμίες μας και κάναμε προσπάθειες σε πέντε επίπεδα παράλληλα με τα μαθήματα που πήραμε από την επιχείρηση Αταλάντα, όχι μόνο για τις τρέχουσες επιχειρήσεις, αλλά και για τις μελλοντικές επιχειρήσεις και όχι μόνο στον τομέα της ναυτικής συνεργασίας, αλλά και στον τομέα των αεροπορικών. Σε επίπεδο πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν μια συνολική προσπάθεια βελτίωσης της ικανότητας που έχουμε και στον τομέα της πληροφόρησης χρησιμοποιώντας συστήματα αεροσκαφών χωρίς πιλότο, χωρίς μη επανδρομένων αεροσκαφών. Υπάρχει επίσης και δυνατότητα βελτίωσης της συνεργασίας ανάμεσα στα στρατιωτικά και τα πολιτικά μέσα. Αυτά δεν είναι θέματα που μπορούν να είναι χρήσιμα μόνο στις εξελίξεις στο στρατιωτικό τομέα, αλλά σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες της γραμματείας που ασχολούνται με θέματα πολιτικά, μη στρατιωτικά εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς καμιά φορά δημιουργούνται επικαλύψεις και αυτό επιβαρύνει οικονομικά τη λειτουργία των συστημάτων. Δύο τελευταία λόγια για τις εταιρικέ σχέσεις, σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Θα ήθελα, δεν θα ήθελα να εστιαστώ στη πολιτική ε, διάσταση, γιατί υπάρχουν κάποια πολιτικά ζητήματα τα οποία είναι γνωστά. Ωστόσο, στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουμε, θα ήθελα να πω στο δικό μου επίπεδο και με τις δικές μου επαφές που έχω με τον ΝΑΤΟ, οι επαφές ε, με τον ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Ανέφερα για την επιχείρηση Ταλάντα, όπου έχουμε πολύ καλό μόντους operandi με τον ΝΑΤΟ, αλλά και με άλλες στρατιωτικές οργανώσεις. Η επιχείρηση Βερολίνο ΣΥΝ συνεργάζονται επίσης πολύ καλά με την επιχείρηση Άλτεα στην Βοσνία και το προσωπικό μου, το επιτελείο μου συναντιέται τακτικά με το επιτελείο του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουμε ότι το έργο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, αλληλοεπικαλύπτεται με το έργο του ΝΑΤΟ. Και αυτό το κάνουμε προκειμένου να ε, μοχλεύσουμε το έργο της άλλης οργάνωσης πάντα έχοντα κατά νου ότι θα πρέπει να διατηρηθεί φυσικά η αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στις ε, αντίστοιχε όργανώσει και φυσικά του σεβασμού των πολιτικών ε, περιορισμών. Η σχέση λοιπόν σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι πολύ καλή με τους δεδομένους περιορισμούς. Ε, αν θα μπορούσε να είναι καλύτερη η σχέση αυτή, φυσικά θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Θα σα το πω με πάσα ειλικρίνεια. Τα προβλήματα όμω δεν είναι σε επιχειρησιακό επίπεδο. Το πρόβλημα έγκυται ε, σε πολιτικό επίπεδο και άρα δεν αποτελεί δικό μου, δική μου ευθύνη. Η σχέση τώρα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα. Θα έλεγα ότι και αυτή έχει βελτιωθεί πολύ. Κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι τα επιτελεία στις ε, δύο οργανώσεις θέλουν να προωθήσουν, αν θέλετε, ζητήματα ιδιοκτησίας ε, των ε, project και θεωρώ ότι αυτό είναι μάλλον αυτονόητο, γιατί πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν δουλέψει σκληρά για τα project αυτά και θα πρέπει να σας πω ότι η σχέση μου, η σχέση μεταξύ του επιτελείου μας και του επιτελείου του Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Άμυνας είναι καλύτερη από κάθε άλλη στιγμή τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό δεν το θεωρώ δική μου προσωπική νίκη, αλλά θέλω να πω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη τώρα. Κοιτώντας την επιχείρηση Τσάντ. Πρέπει να σας πω ότι από στρατιωτικής απόψης και σε επιχειρησιακό επίπεδο τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η συνεργασία ήταν εξαιρετικά καλή. Φυσικομικές δυσκολίες, υπήρχαν ε, χρηματοοικονομικές ε, δυσκολίες και αυτό αποτέλεσε μέγα εμπόδιο, αλλά σε στρατιωτικό επίπεδο υπήρχε καλή συνεργασία και όλα πήγαν καλά. Φυσικά δεν μας ικανοποιεί αυτό μόνο και θα πρέπει να διδαχτούμε από τα παθήματα του παρελθόντος και την προηγούμενη εβδομάδα είχα ακόμα εκπροσώπους που ήρθαν να κάνουν ε, ελέγχους στη γραμματεία για να διασφαλίσει ότι είχαμε μάθει πραγματικά από τα παθήματα του Τσάντ. Και μια τελευταία κουβέντα τώρα, πρωτού σταματήσω για κάποια θεσμικά ζητήματα, κάποια θέματα διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχετικό προσωπικό έχει, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει περιοριστεί, το οποίο μπορεί να σας προκαλέσει έκπληξη. Όταν ήρθα, όταν ξεκίνησα, ήταν περίπου στη 200. Μετά είδαμε τι έγινε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και είπαμε τα παθήματα του Βίσμπαντ αποκαλέστηκαν αυτά τα παθήματα όπου λάβαμε εντολή για τον καλύτερο και πιο πρώιμο σχεδιασμό των ε, project αυτών και ενισχύθηκε το επιτελείο μας με 10 αξιωματικούς και κάναμε μία αναδιοργάνωση του στρατιωτικού επιτελείου προκειμένου να είμαστε έτοιμοι και να κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό των ε, επιχειρήσεων. Αυτό πήγε πολύ καλά και νομίζω ότι η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι σε κάποια από τα σχέδια που καταστρώθηκαν για το Τσάντ, για την Αταλάντα και για την ε, εκπαιδευτική αποστολή στην ε, Σομαλία έχει αποδεχτεί πραγματικά αυτή η προστιθέμενη αξία και καταφέραμε να ενισχύσουμε και την ε, πολιτική διάσταση του σχεδιασμού αυτού. Η τελευταία εξέλιξη, όπως ξέρετε, είναι η Η ανάπτυξη του CSPD υπό την, την ηγεσία της κυρίας Παντού, 14 μέλη του Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δοθεί μεγαλύτερη στρατιωτική διάσταση στο CNPD και αυτό έχει αυξήσει την αριθμητική ισχύ του Ευρωπαϊκού Επιτελείου και πάλι θα πρέπει να σας πω ότι κάναμε κάποιες θυσίες σε κάποιους τομείς, αλλά δεν θυσιάσαμε, πρέπει να σας πω, ε, την οργανωτική μας δυνατότητα βάσει των μαθημάτων του Βίσμπάντεν, όπως τα αποκαλούμε. Και θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε την κρίσιμη μάζα για να εκπληρώνουμε την εντολή μας όταν χρειάζεται, αλλά παράλληλα θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τον αντίκτυπο της Διεύθυνσης ε, Διαχείρισης Κρίσεων που έχει αναλάβει κάποιες ε, από τις ε, αρμοδιότητες. Θα πρέπει να δούμε όμως αν σε έξι μήνες το επιτελείο είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του και φυσικά η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Υπήρξε αρχικά ένα σχέδιο να ενταχθούμε κι εμείς στην υπηρεσία αυτή. Αυτό είναι το σχέδιο, δεν έχει αλλάξει. Όπως ξέρετε είπα ότι ε, εκπρόσωπος αφιερώνει μεγάλο τμήμα των προσπάθειών της για την διοργάνωση και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων της εξωτερικής υπηρεσίας και θα πρέπει να σας πω ότι συμμετέχουμε ιδιαίτερα στα πλαίσια του σχεδίου αυτού και θα σας παρουσιάσουμε τα σχέδια αυτά συντόμως. Thank you, General. Θα σας ευχαριστώ και τώρα να ακούσουμε τις ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Καταρχάς να ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Ο συνάδελφος Γκάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντιστράφηγε Λίκη μετά τα τρία χρόνια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τη θητεία σας. Καταρχάς για το γεγονός ότι πολλές φορές ήρθατε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και για την πάντα επαγγελματική σας ε, και άξια παρουσίαση των ε, εξελίξεων. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι πραγματικά πάντα επωφελήθηκαν ιδιαίτερα και επηρεάστηκαν και οι πολιτικές μας ε, αποφάσεις. Ενδιαφέρον ήταν ότι ακούσαμε ότι στα πλαίσια της ε, Αταλάντα είναι πολυεθνική η συνεργασία που έχει εγκαθιδρυθεί και λειτουργεί καλά οι διαφορετικές ε, οργανώσεις, τρεις, ίσως και αν προσταθεί και εκείνα τέσσερις να είναι στον αριθμό, συνεργάζονται σωστά. Είπατε επίσης ότι προσέχουμε ιδιαίτερα να μην υπάρχουν ε, επικαλύψεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Αν σε μια επιχείρηση συμμετέχει στη φάση της διοργάνωσης ε, Τη οργάνωση και του σχεδιασμού και των ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται ούτω ή άλλω ε, για επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Ίσως αυτό θα πρέπει να διοργανωθεί διαφορετικά το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Μπόντ. Ίσως θα χρειαστεί να έχουμε σε διαφορετικό σκέλος την, ε, το σχεδιασμό και την εφαρμογή. Τώρα που αποχωρείτε από τη θέση σας και έχετε πιο μεγάλη ελευθερία έκφρασης, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι δική σας άποψη. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ούτως ή άλλως πρόκειται για καλή συνεργασία και άρα δεν χρειάζεται περαιτέρω βήματα. Μία άλλη ερώτηση για κάτι το οποίο δεν θίξατε, αλλά που μας απασχολεί ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή ε, πολιτική σκηνή. Έχουμε φιλόδοξα σχέδια σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές μας και το 2004 έχουμε ορίσει μάλλον ε, τους ε, σχετικά ε, κεφάλαια 2004-2010. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα για την ενίσχυση των ικανοτήτων μας και τη σχετική διακήρυξη και δήλωση του 2008 Πού θεωρείτε λοιπόν σε σχέση με αυτή τη δήλωση ότι έχουμε πετύχει και πού απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ επαγγελματική παρουσίασή σας και την πάρα πολύ ενημερωτική επίσης παρουσίαση και θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι επενήσατε και τους ε, αντι, αντιπάλους σας στο παιχνίδι του με τις επόμενες δεκές. και να σας ε, ευχηθώ καλή επιτυχία στην ε, νέο σας ρόλα. Ίσως πιστεύετε ότι η πολιτική ήταν κάτι καλύτερο Θα με ενδιαφέρα να μου πείτε το εξής. Πόσο ποσοστό της Αταλάντα βασίζεται στον καλό σχεδιασμό σας για την, ε, ε, την καλή σας οργάνωση και την καλή παρακολούθηση του γινόταν στην περιοχή της Σομαλίας. Επίσης, είπατε ότι ασχολείστε με την κατάρτεση των μελλοντικών στρατιωτών στην Σομαλία. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι μισό με αυτό που κάνετε εσείς. Το άλλο μισό το διαδραματίζουν τα θεσμικά ε, οι θεσμοί αν θέλετε, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν σωστά τους στρατιώτες και το προσωπικό που εσείς καταρτίζετε στη Σομαλία. Επίσης, όταν καταδικάζονται οι Σομαλοί, πού πηγαίνουν, πού φυλακίζονται ενδεχομένως για να εκτίσουν την ποινή τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Αντιστράτηγε, νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά από σας. Λυπούμε που εγκαταλείπετε τον ε, παρόντα καθηκοντά σας. Εσείς να μπορούσατε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο τώρα. Το χόμπι σας μήπως θα ήταν να ασχοληθείτε με την ε, πολιτική ή να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Πριν όμως πάρετε μια τέτοια απόφαση να φύγετε, οι παρατηρήσεις που κάνατε με κάνουν να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβω καλύτερα τα πράγματα. Με την επιχείρηση Αταλάντα. Εσείς κρίνετε ότι μέχρι τώρα ως επιχείρηση ήταν επιτυχής. Έχω δύο ερωτήσεις σχετικά. Σε σχέση με την συνεργασία την οποία αναφέρατε με χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, που προφανώς ε, συμμετείχαν θετικά. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άλλα καθήκοντα για τα οποία τέτοιου είδους συνεργασία με τέτοιες χώρες θα ήταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση μία από τις επιλογές δεύτερον. Όσον αφορά το ρόλο του ε, πολιτικού σκέλους της συνεργασίας και όλων αυτών οι οποίοι συμμετέχουν από πολιτική σκοπιά. Ποιος είναι ο ρόλος τους στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η επόμενη μου παρατήρηση αφορά την αποστολή Ιούσον. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η συνεισφορά των διαφόρων κρατών μελών σε αυτή την αποστολή. Μπορείτε να μας ε, απαριθμίσετε κάποιες χώρες. Τρίτον, ποιες προφυλάξεις και μέτρα παίρνουμε κατά του κινδύνου απόσυρσης κάποιων ή αποχώρησης. Ίσως καταρτίζουμε εμείς ε, στρατιώτες κάπου οι οποίοι κάποια στιγμή θα πάνε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως καταρτισμένοι σε κάποιον πολέμαρχο σε κάποιες χώρες επικίνδυνες. Επίσης, πώς μετράτε την επιτυχία των επιχειρήσεών σας. Επίσης, για την συνεργασία με τον ΝΑΤΟ θα σημειώσατε ότι στην στρατιωτική σχολή τον Ιανουάριο ο, η Χίλαρη Κλίντον όταν αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή ε, ασφάλεια δεν αναφέρθηκε καθόλου στην ε, ΚΕΠΑ. Πιστεύετε εσείς από τη μεριά του ΝΑΤΟ ο ρόλος της ΚΕΠΑ υποβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο ή συνειδητοποιεί το ΝΑΤΟ το ρόλο τον οποίο εμείς μπορούμε να διαδραπεντήσουμε στα πλαίσια αυτής της πολιτικής. Κύριε Στάνοκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιστράτη Γελική για την Αταλάντα. Ξέρω ότι ε, κάνατε νομικά στο Κέμπριτς πριν να ασχοληθείτε με στρατιωτικά θέματα. Θέλω να μας πείτε κάποια πράγματα για την ε, νομική βάση την οποία εμείς βασιζόμαστε για να μπορέσουμε να συλλάβουμε ή να αναχαιτήσουμε κάποιους πειρατές. Και τι γίνεται με την ε, ε, Κένια. Είπατε ότι στην Κένια δικάζονται το δικαστικό σώμα της Κένιας Πολλές φορές έχει κάνει στις δικές μας χώρες τις ε, σπουδές του. Πώς συμπεριφέρονται. Επίσης, κάποια χρήματα τα οποία καταβάλλονται ε, από ε, κάποιους πώς χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται για, από την ε, Τζιχάν. δεδομένης της μεγάλης σημασίας της ε, του, της περιοχής του κέρατος της Αφρικής, τι πιστεύετε ότι ε, μπορεί να γίνει επίσης. Δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος για κάτι το οποίο είπατε. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε κάποιους από εμά που έχουν κάποιο σκεπτικισμό όσον αφορά την ε, ΚΕΠΑ ότι κάποιες ε, ε, χώρες όπως η Ινδία συμμετέχουν ενεργά σε κάποιες συμμαχικές ναυτικές επιχειρήσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε ή οι οποίες αναλαμβάνονται υπό την από, την, από το ΝΑΤΟ, γίνονται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και αποτελούν σε θέματα συνεργασίας μία προστιθέμενη αξία για μας. Επίσης, είδα ο, στο, στο βιογραφικό σας ότι μαθαίνετε και ξένες γλώσσες. Πρόσφατα ποιες γλώσσες μάθηκε, ποιες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε εκτός από την αγγλικά. Ποια είναι η δεύτερη γλώσσα την οποία μάθατε εσείς. Επίσης μπορείτε να μας πείτε επισήμως ή ανεπισήμως πότε συναντάτε, συναντάτε τον Σασέρ, τον ε, Γενικό Διοικητή ε, του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας πω ευχαριστώ, αλλά επειδή είμαι ευγενής θα πω ευχαριστώ. Πολύ πλούσιο το μενού. Ας αρχίσω με την πρώτη παρατήρηση που αφορούσε την άποψή μου για το ε, τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλε μου τις παρατηρήσει είναι κάτι που θέλω να το επαναλάβω ότι είναι αληθέ ότι όλοι οι Βρετανοί όταν γεννούνται είναι ευρωσκεπτικιστέ, το έχουν στα γονίδια. Και εγώ είμαι ένας από αυτού. Είμαι ευρωσκεπτικιστή και το δηλώνω. Για πολλούς λόγους και από τότε που είμαι εδώ στις Βρυξέλλες εδώ και τρία χρόνια γίνομαι όλο και λιγότερο ευρωσκεπτικιστής και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους μπορεί κανείς να είναι ευρωσκεπτής αλλά στον τομέα της ΚΕΠΑ, στον τομέα τον δικό μου είναι το στον οποίο μπορώ να εκφράσω τον λιγότερο σκεπτικισμό ε, σήμερα και θα σας εξηγήσω για ποιους λόγους. Ας αρχίσουμε όμως με τις ε, με τη Γενικό Επιτελείο το Επιχειρησιακό, όπου σχεδιάζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και εδώ πρέπει να έχουμε ε, πάρα πολύ καλό επιχειρησιακό επιτελείο για να το κάνουμε αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικό το επιτελείο μας. Έχουμε το SHAPE για το Βερολίνο ΣΥΝ, Έχουμε το Πόσταμ, το Northwood που πραγματικά έχουν αποδείξει ότι αξίζουν. Όλοι οι εγκαταστάσεις με το προσωπικό τους είναι εξαιρετικές. Υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν κοστίζουν πολύ. Πολύ καλά επανδρομένος. Δεν θέλω να επικρίνω καμία από αυτές τις τρεις εγκαταστάσεις που ανέφερα, τρία αυτά επιταλεία. Η επιχειρήση Αταλάντα πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, αλλά ηγείται το επιτελείο του Northwood. Δεδομένου ότι είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα επιτελείο για ναυτικές επιχειρήσεις, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές και πολύ χρήσιμες και επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ανακυκλώνουν και άτομα τα οποία πηγαίνουν εκεί στο στρατηγείο εκεί και να βλέπουν στην πράξη καθημερινά πώς ε, λειτουργεί μια τέτοιου είδους οργάνωση. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ προστιθέμενη αξία και τα επιτελεία λειτουργούν πολύ σωστά. Τώρα, τι γίνεται Ε, για να το πω αγγλικά, κάτι που, δεν λειτουργεί, κάτι που λειτουργεί σωστά, τι κάνουμε για να το κάνουμε καλύτερα να το διορθώσουμε. Κάνουμε ανάλυση. Διότι, εάν θέλετε να ιδρύσετε ένα στρατηγείο, θα πρέπει να ξέρετε πρώτα απ' όλα αν έχετε την εγκατάσταση, αν μπορείτε να το επανδρώσετε, πόσο μεγάλο θα είναι το στρατηγείο, και ορισμένοι σας, λέει ότι, ε, σας λένε ότι μπορείτε να έχετε 40, 60, 100 άτομα αλλά λέγεται να ασχοληθείτε με μία ή δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ίσως θα πρέπει να το επανδρώσετε με περισσότερα άτομα. Όταν όμως έχετε πλήρη στρατηγία, με πλήρως επανδρωμένα, με καταρτισμένα άτομα, τα σωστά άτομα στη σωστή θέση που μπορούν να ανταποκριθούν ε, ταχύτατα τα αιτήματα, όσο μεγάλο και να είναι, με 200 άτομα, 400 άτομα, στο οποία μπορείτε να έχετε προσωπικό το οποίο να έρχεται από κάπου αλλού παρά τις ε, οικονομικές ε, δυσκολίες που υπάρχουν παντού μπορείτε να λειτουργήσετε. Και εκεί πολλές φορές που δεν υπάρχει ε, αρκετό προσωπικό ΝΑΤΟ, μπορείτε να έχετε προσωπικό Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχετε όλες αυτές τις δυνατότητες συμπληρώνοντας η μεν δε. Τώρα, μας ρωτάει ο κύριος Τάνοκ, η... και από πόσο χρήσιμη είναι. Θα ήθελα να πω το εξή. Σωστά θέσετε το θέμα. Η ΚΕΠΑ πληρώνει ένα κενό στην αγορά, αν θέλετε. Αυτό το έχει αποδείξει πολλές φορές. Φερρυπίν. Η αποστολή στο Τσάντ δεν θα μπορούσε να είχε γίνει μόνο από το ΝΑΤΟ. Δεν θα είχε γίνει αυτό αποδεκτό ε, για τις κυβερνήσεις των κρατών της Κεντρικής Αφρικής μόνον από το ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν η διεθνής κοινωνία είπε πρέπει να κάνουμε κάτι στο Τσάντ, διαφορετικά θα, η κατάσταση τύπου Νταρφούρ θα επεκταθεί πολύ και θα έχουμε πολιτικό και ανθρωπιστικό πρόβλημα. Άρα είπαμε ότι θα πρέπει προληπτικά να κάνουμε κάτι, να αναλάβουμε δράση και η διεθνής κοινότητα, ακόμη και τα Ηνωμένα, ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείες, ενθάρρυναν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει κάποιο ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Διότι χρειαζόταν κάποιο κάτι να κάνει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία πολιτική ε, ομπρέλα, αν θέλετε, έχει ε, την πολιτική κατάλληλη ηγεσία και έχει και το στρατιωτικό περιορισμένο προσωπικό που έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, το μικρό προσωπικό των 180 περίπου ατόμων για μισό εκατομμύριο Ευρωπαίων, αλλά εν πάση περιπτώσει 177 άτομα ήταν ικανά να ηγηθούν των επιχειρήσεων στο τσάντ και να πληρώσουν αυτό το κενό που υπήρχε στην αγορά, όπω είπα στην αρχή. Τώρα, αν θα έπρεπε να είναι επιχείρηση ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πω ότι σε επίπεδο διοίκησης, επειδή υπήρχε το επιτελείο δεν κόστησε ούτε ένα φράγκο παραπάνω η όλη αυτή η επιχείρηση στο ΝΑΤΟ. Κόστισε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 114 άτομα περισσότερα, αλλά 114 περισσότερα άτομα σε όλη την Ευρώπη να, για να συμμετέχουν σε μία ναυτική επιχείρηση είναι πολύ φτηνό αν θέλετε. Πολύ φτηνό. είναι είναι σαν την EasyJet. Εν πάση περιπτώσει, η οργάνωση, γενικότερα η ομπρέλα που σας είπε αυτή, η οποία προσέφερε αυτή την προστιθέμενη αξία και σε τέτοιου είδου επιχειρήσει διευκολύνεται και η συνεργασία με άλλε δυνάμει όπω η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία. Και σα λέγω ότι εάν ε, όλα είχαν γίνει αποκλειστικά μόνο από άλλε οργανώσει και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη εξοπλισμό. Δεν θέλω να ε, πω τίποτε κατά του ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να σας πω ότι με την ε, παρουσία του ΝΑΤΟ και με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες που θέλησαν να συμμετάσχουν δώσαν να συμμετάσχουν και το γεγονός ότι το τι κάνει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επικάλυψη αλλά ως συμπληρωματικές δράσεις. Αυτό θα έλεγα αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο φέρει μία προστιθέμενη αξία εξαιρετική και σε πολύ, με πολύ χαμηλό κόστος, με 114 μόνο συμπληρωματικά άτομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ σωστό. Τώρα, αν χρειαζόμαστε εδώ πέρα στις Βρυξέλλες να έχουμε ένα επιτελείο πιο καλά επιδρομένο, πιο μεγάλο, θα χρειαστεί χρόνος για να κρίνουμε αν χρειάζεται κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι θα πρέπει πριν να ληφθεί μια τέτοια απόφαση να ε, εξετάσουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως να κάνουμε μια εξαιρετική ανάλυση. Και ένα μεγάλο μέρος της ανάλυσης θα είναι αυτή η συνολική προσέγγιση που θέλουμε να έχουμε. Ποιο είναι το επίπεδο των δικών μας φιλοδοξιών για αυτή την ε, σφαιρική προσέγγιση. Ξέρουμε τι σημαίνει μία επιχείρηση πολιτικό-στρατιωτική. Ε, θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο ε, ενσωματωμένο και υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Στην γραμματεία, στο ΝΑΤΟ, στα κράτη-μέλη πάτε σε τα σεμινάρια και σα λένε ότι θέλουμε να έχουμε δύο διαφορετικά επιτελεία, το πολιτικό σκέλος και το στρατιωτικό χωριστά. Ο καθένα έχει τη δική του κουλτούρα και αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη και τα συντάγματα κάποιων χωρών το προβλέπουν. Πριν αρχίσουμε λοιπόν να βιαζόμαστε και να θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο επιτελείο, θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το επίπεδο των φιλοδοξιών, για το ποιο είναι ο στόχος τον οποίο θέλουμε και αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι... Um, Η συζήτηση λοιπόν σήμερα είναι κατά πόσο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους στόχους που αναφέρατε, κατά πόσο θα πρέπει να τους ξαναγράψουμε. Κανείς δεν έχει εκβαστεί ακόμα, αλλά να σας πω προσωπικά τη δική μου τοποθέτηση, μια και αποχωρώ, μπορώ να σας δώσω την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι ναι, θα πρέπει να τους ε, αναθεωρήσουμε, αλλά τη σωστή χρονική στιγμή. Σήμερα, στην παρούσα φάση, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες ανατρεπτική. Να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Δεν έχει νόημα όταν το πλαίσιο μετατρέπεται και αλλοιώνεται να θέσουμε νέους στόχους και θα πρέπει να σκεφτούμε τρία πράγματα. Ποιο είναι η μελλοντική μορφή των συγκρούσεων, αυτό να το λάβουμε υπόψη. Κοιτώντα και τους στρατούς, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι κάποιοι αλλάζουν ε, οργάνωση. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 10-20 χρόνια. Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο που μας απασχολεί. Θα χρειαστούμε πολλά σκάφη, αεροσκάφη, πολεμικά σκάφη και το καθεξής. Τέτοια θέματα θα πρέπει να σκεφτούμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης τι μάθαμε από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τα Βαλκάνια. Για να δούμε πού μας οδηγούν τα συμπεράσματα, τα πορίσματα, τι θα χρειαστούμε στο μέλλον. Και αυτό μας ξαναφέρνει στην συνεκτική, ενιαία προσέγγιση. Πόσο θα πρέπει να συντονίζεται το σκέλος, το στοχευτικό και το πολιτικό. Αυτό αποτελεί λοιπόν ένα παράγοντα, μία συνιστόσα. Κατά δεύτερον, βρισκόμαστε σε μία δύσκολη οικονομική κατάσταση και Αυτό θα επηρεάσει και τον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές επενδύσεις. Είναι λοιπόν κατά ηλεκτρονική στιγμή να θέσουμε νέους στόχους. Και άλλο ένα σκέλος που είναι η στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ. Να δούμε ποια θα είναι η φιλοδοξία του ΝΑΤΟ, γιατί αν υπάρχει συμπληρωματικότητα, ας διαμορφωθεί με το σωστό τρόπο, προκειμένου να υπάρξει εγγύηση τη συμπληρωματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο το ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντω υπάρχουν και άλλοι παράγοντε. Τι γίνεται στον ΟΗΕ που βρίσκεται σε φάση μεταρρύθμιση. Ενώ λοιπόν η διεθνή κοινότητα βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωση, το να αναθεωρήσουμε του στόχου αυτού τώρα ίσω θα ήταν ε, λίγο βεβαιασμένο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο δεν βλέπω να υπάρχουν οποιασδήποτε ενδείξει ε, δραματικών ε, αλλαγών, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξει για μικρές βελτιώσει σε κάποιου συγκεκριμένου τομεί. και νομίζω ότι ακόμα και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αναγκάζουν κάποιους ανθρώπους να αναδιοργανώσουν, να ομαδοποιήσουν αν θέλετε τις αρμοδιότητέ τους στρατηγικές, στρατηγικές αερομεταφορές, αεροπλανοφόρα, ακόμα και οι πολεμικοί σχηματισμοί είναι αντικείμενο μεταρρύθμισης. Για την αξία των πληροφοριών για την Αταλάντα. Είναι χρήσιμες φυσικά οι διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά. Το σύστημα πάντως λειτουργεί, μαζεύει πληροφορίες, είναι λειτουργικές αυτές τις πληροφορίες και ε, ε, είναι κάτι το οποίο είναι αξιόλογο. Τον προηγούμενο μήνα συλλάβαμε 60 περίπου ε, πειρατές, καταστρέψαμε 11 σκάφη και αυτό το πετύχαμε μέσω των πληροφοριών τις οποίες συλλέξαμε και μέσω επίσης των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. Υπάρχει νομίζω μια καλή προσπάθεια συνεργασίας και σε επίπεδο τακτικό στα πλαίσια της διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Και η κατανομή πληροφοριών έτσι ώστε να μπορέσουν και άλλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τους στόχους τους οποίους εμείς έχουμε εντοπίσει είναι κάτι το θετικό. Για την εκπαίδευση των Σομαλών θα συμφωνήσω με την παρατήρηση ότι η Αταλάντα από τη μία και από την άλλη η προσπάθεια εκπαίδευσης των Σομαλών δεν θα λύσει το πρόβλημα της Σομαλίας. Ακόμα και αν λυθεί το πρόβλημα των πειρατών, ε, το πρόβλημα της Σομαλίας είναι μακροπρόθεσμο και σοβαρό. Αλλά δεν θα σχολιάσω εγώ περισσότερο τον τομέα αυτό. Υπάρχει όμως ένας πολύ μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων για τη Σομαλία που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίδει και έχει προσημειώσει πάρα πολλά χρήματα για τη Σομαλία, 87 συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία έχουν σαν στόχο τη Σομαλία. Συνεπώς, ο συνολικός τρόπος αντιμετώπισης του σομαλικού προβλήματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητος, αλλά βέβαια είναι και κάτι το οποίο θα πάρει πολύ χρόνο. Λοιπόν, το chainsawing είναι κάτι το οποίο σαν δραστηριότητα είναι χρήσιμο και για τους πολιτικούς και για τους στρατιωτικούς. Λοιπόν, για τα μαθήματα που πήραμε από την Ανταλάντα σε συνεργασία με τους ε, οι, οι, ε, Κινέζους, ε, Ινδούς κτλ και ίσως να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες αυτές για να καλέσουμε και άλλες χώρες να πάρουν μέρος σε άλλες τις επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ στο μέλλον. Αυτό όμως που γίνεται στην Αταλάντα δεν είναι καινούριο. Δεν έχω εγώ τον κατάλογο όλων των χωρών, όταν ήμουν όμως υπεύθυνο για τη U4 στη Βοσνία, υπήρχαν σχεδόν 40 χώρες οι οποίες είχαν στείλει στρατό στη U4. και οι περισσότερες ε, φυσικά ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του ΝΑΤΟ, αλλά πολλές ήταν από μακρινές περιοχές, Λατινική Αμερική κτλ. Το να ανοίξουν λοιπόν οι ενέργειες, οι δραστηριότητες συγγνώμη, της ΚΕΠΑ σε ξένες δυνάμεις, σε μακρινές χώρες, αυτό είναι παλιά πρακτική. Ε, αυτό που δεν συζητάμε πάρα πολύ, καλά είναι η, η ρωσική συνεισφορά στην επιχείρηση στο Τσάβε. Είναι τα, ελικόπτερα βαρέων μεταφορών που μας διέθεσαν οι Ρώσοι, όπως επίσης και τα ελικόπτερα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την διακομιδή των ασθενών και τραυματιών. Ε, η συνεισφορά των Ρώσων δηλαδή στο Τσάδι ήταν σημαντική. Τώρα, ο κίνδυνος ε, λιποταξιών από την δύναμη ε, εκπαιδευομένων Σομαλών. Ε, είναι αλήθεια ότι μπορεί να πάνε σε αυτόν που τους δίνει τα περισσότερα. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος. Ε, μία από τις προϋποθέσεις ε, στις οποίες επιμένουν τα κράτη-μέλη για την προσπάθεια αυτή την εκπαιδευτική είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο και να γίνει κάθε βήμα για να αποτραπούν οι λιποταξίες. Κάποια από τα μέτρα αυτά είναι τα εξής. Πρώτον, θα πληρώνονται ε, λίγο φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Δεν ξέρω και δεν θα πω από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε χρηματοδοτούν αυτό το... Secondly, the salaries, once they return to Mogadishu, uh, the US have αυτό το χαρτζηλίκι σε εισαγωγικά το οποίο θα τους δίνουμε. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξει μια δυνατότητα κάλυψης κατά 50% των χρημάτων που θα δοθούν για την πληρωμή των μισθών των ε, μελών των ε, δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας. Πρέπει να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε και το υπόλοιπο 50%. Υπάρχει αισιοδοξία όμως γιατί στη συνάντηση των δωρητριών χωρών που έγινε στις Βρυξέλλες πριν από αρκετούς μήνες, λιγότερο από ένα χρόνο, είπαμε ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή θα μπορούσε θα έλεγα ο προσανατολισμός τους να αλλάξει έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ε, των σομαλικών ε, ε, ενόπλων δυνάμεων. Ένα δεύτερο θέμα είναι αν οι Σομαλοί θα πάρουν αυτά τα χρήματα βέβαια, είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχει ο κίνδυνος να στείλουμε στο Μογκαντήσου χρήματα και όποιος θέλει να πάει στη Σομαλία και να μοιράζει τα χρήματα αυτά στα γραφεία ή στο δρόμο, στους Σομαλούς να μου το πει να τον στείλω γιατί πρέπει να είναι πολύ γενναίος και ανόητος για να το κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να δοθούν σε αυτούς για τους οποίους προορίζονται. και η Cooper έχει ήδη αναλάβει μια διαδικασία η οποία μέχρι τώρα φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική και τα χρήματα θα φτάσουν σε αυτούς για τους οποίους προορίζονται. Δύο ακόμα πράγματα. Πρώτον, οι δυνάμεις ασφαλείας της Ομαλίας όταν επιστρέψουν στην χώρα τους θα ελέγχονται από την επιχείρηση Έμεσον και ένα τμήμα της εκπαίδευσης το οποίο θα λάβουν στο τέλος μάλλον της διαδικασίας ε, θα έχουν τους λεγόμενους, ε, όχι ηγέτες τους, αλλά τους μέντορές τους θα έλεγα, για να τους ελέγχουν και στην ουσία θα συνδεθούν μαζί τους έτσι ώστε όταν επιστρέψουν στο Μογκαντήσου να υπάρχει μια ουσιαστική επίβλεψη της συμπεριφοράς αυτών των στρατιωτικών δυνάμεων. Θα υπάρξουν δύο επίσης διαδικασίες ελέγχου. Καταρχάς οι νεοσύλλεκτοι στο Μογκαντήσου θα ελεγχθούν από την Έμεσον και τώρα κάποιοι θα πούν είναι αποτελεσματικό αυτό. Αυτό θα το ρωτήσετε στους ε, εκπροσώπους της κυβέρνησης της Ουγκάντα. Βέβαια η Έμεσον δεν είναι μόνο η Ουγκάντα αλλά παρόλα αυτά έχουν εμπλακεί ιδιαίτερα η, η, κυβέρνηση της Ουγγάντα και μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στη Σομαλία μόνο εφόσον οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας αυτής επιτέλους αποκτήσουν την ικανότητα να ελέγχουν την κατάσταση αυτή. Λοιπόν, ε, υπάρχουν κίνητρα εδώ και για τους ε, εκπροσώπους της κυβέρνησης της Ουγγάντα να κάνουν σωστές διαδικασίες ελέγχου. Θα υπάρξει ένας δεύτερος έλεγχος των δυνάμεων αυτών όταν φτάσουν στην Ουγγάντα, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ανάμεσα σε άλλα ότι δεν εκπαιδεύουμε κόσμο παραβιάζοντας, αν θέλετε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρθηκα στι Ηνωμένε Πολιτείε ήδη. Η συνεργασία ανάμεσα στην ΚΕΠΑ και το ΝΑΤΟ είναι ένα θέμα. Υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας ΚΕΠΑ και ΙΠΑ. Με ακούσατε να λέω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πληρώνουν του χαρτζιλίκη των σώμαλών εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής εκπαίδευσης και όχι μόνον αυτό, αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα δώσουν και τον εξοπλισμό που απαιτείται και θα χρηματοδοτήσουν και κάποιες από τις αποδομές, θα καλύψουν το κόστος το οποίο θα προκαλέσει η εκπαίδευση αυτή. Αυτό δεν θα γίνει μονομερός, γίνεται σε στενή συνεργασία με εμά. Έγινε μια συνάντηση στη Καμπάλα ε, πριν δύο εβδομάδες έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένε Πολιτείες και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του Ουγγάντα και άλλου εταίρους. Είναι η πρώτη μορφή άμεσης συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα, το νομικό κενό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δίωξη των πειρατών. Δεν είναι αλήθεια να μιλάμε για νομικό κενό. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χαρακτηρίζονται από ένα τέτοιο νομικό κενό. Υπάρχει όμως μια έλλειψη επιθυμίας να φέρουμε εδώ τους Σομαλούς και να τους δικάσουμε. Και ε, γιατί έτσι θα αυξήσουμε τη διασφορά των Σομαλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω λίγο έμεσα. Δεν είναι αλήθεια να λέμε επίσης ότι οι Κενιάτες δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα. Η ίσα ίσα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τα μέσα, τα οικονομικά, στο δικαστικό και σοφρονιστικό σύστημα της Κένια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και οι πειρατέ οι οποίοι διώκονται και φυλακίζονται στην Κένια να παραμείνουν στη φυλακή εκεί και οι φυλακές της Κένια να είναι στα σωστά επίπεδα. τι παίρνουν ε, ε, οι, οι ομάδες, οι ανεξέλεγκτες της Σομαλίας, οι ένοπλες, από τα χρήματα και τα λίτρα τα οποία εισπράττουν οι πειρατές. Έχουν υπάρξει ε, πάρα πολλές παραπλανητικές δηλώσεις θα έλεγα. Έχουν δημοσιευθεί κάποιες, κάποια στοιχεία θα έλεγα από μη κυβερνητικέ οργανώσεις στα μέσα ενημέρωσης που διαψεύδουν τις επίσημες δηλώσεις των χωρών της περιοχής. Και από ό,τι φαίνεται κάποιες ομάδες ένοπλες της Σομαλίας ε, παίρνουν ένα κομμάτι των λίτρων τα οποία εισπράττουν οι πειρατές. Αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα την ανακριτική ε, να, να, να αποδείξουμε ή να διαψεύσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς για το Πούτλαντ και το Σόμαλιλαντ, τις περιοχές αυτές η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχύει την κυβέρνηση της Σομαλίας και να μπορέσει το Μογκαντήσου να ελέγξει και την υπόλοιπη χώρα. Το Πούντλαντ και το Σόμαλιλαντ. Έχει υπάρξει όμως υποστήριξη άμεση των αρχών των τοπικών στο Πούντλαντ και στο Σόμαλιλαντ. Σε στρατιωτικό επίπεδο έχουμε επαφές μαζί τους πάρα πολύ συχνά στα πλαίσια της επιχείρησης Ανταλάντα βρίσκομαι σκάφη τα οποία είναι ακυβέρνητα στη θάλασσα, κάποια από αυτά είναι αλλιευτικά. Όλα αλλιευτικά είναι βέβαια τα σκάφη αυτά, αλλά δεν έχουν ε, όλα αλλιείς επάνω τα αλλιευτικά σκάφη και δεν υπάρχουν και αλλιείς γυναίκες φυσικά. Κάποιοι από αυτούς είναι σωματέμποροι ουσιαστικά, είναι αλληλείς ανθρώπων ουσιαστικά. Και προσπαθούμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τις αρχές ε, αυτές για να δούμε τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους τους οποίους διασώζουμε στην περιοχή. Κάποια κράτη-μέλη έχουν και συγκεκριμένα προγράμματα εκεί για να βοηθήσουν τη δημιουργία λιμενικών ε, εγκαταστάσεων και υποδομών στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να προστατεύουν την αλία και τα λοιπά για τη γλώσσα. Θα συνεχίσω στα γαλλικά. Θα σας μιλήσω γαλλικά. Donc, euh, pas tout le monde euh, parle français aussi couramment que moi, euh, mais δεν ομιλούν όλοι τόσο σωστά γαλλικά όσο εγώ. αλλά σε καμία περίπτωση δεν ε, θα συνεχίσω να το κάνω γιατί αλλιώς θα καταστρέψω τη γλώσσα του Μολιέρου και συνεχίζει γερμανικά. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσω γερμανικά, εντάξει. Για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ τώρα. Συναντιέμαι με εκπροσώπους του ΝΑΤΟ μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα σε επίσημη, ε, ανεπίσημη βάση με τον τα λοιπά. Οι επαφές λοιπόν είναι τακτικές ε, και συχνές και εμπλέκουν και διάφορες ομάδες, ε, συχνά άτυπες αλλά πάντα ουσιαστικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ θα πρέπει να διακόψουμε στι 7 και 4, λέει ο Πρόεδρο. Θα ζητήσω λοιπόν από του ομιλητέ να τηρήσουν το χρονικό όριο του ενό λεπτού. Και να ξεκινήσουμε με τον Αντιπρόεδρο Λίζεκ. Ευχαριστώ, Αντιστράτηγε, για όλε τι πληροφορίε που μα δώσατε. Θα ήθελα να αναθέσω κάποια ερωτήματα για την Ιταλία. Αλλά νομίζω ότι αρκετά ε, ενδιαφέροντα ερωτήματα και αρκετέ καλέ απαντήσει λάβαμε για την επιχείρηση αυτή. Για την ε, Άλτεα και την ε, αποστολή στη Βοσνία Ζεγοβίνη συναντηθήκαμε με την πριν από κάποιες ημέρε με τον Υπουργό Άμυνα τη Ισπανία και μα είπε ότι υπήρξε σχετική συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Άμυνα. Κάποιοι εξ αυτών ε, αποφάνθηκαν ότι η κατάσταση πλέον έχει σταθεροποιηθεί και μπορεί να τερματιστεί η επιχείρηση, ακόμα και φέτος ακόμα. Συμφωνείτε με αυτή την αισιοδοξία που εκφράστηκε. Η κυρία Γκομές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Αντιτράτηγε. Θα μας πείτε δύο λόγια για την αποστολή ΚΕΠΑ που λαμβάνει η χώρα στη Γουινέα Μπισάου. Ε, σημειώνεται κάποια διαφορά ή όχι. Είναι σημαντικό γιατί είναι στο κατόφλι της ε, Ένωσης και ε, μιλάμε για λαθρεμπόρια των ναρκωτικών και άλλες μορφές εγκλήματο. Μία δεύτερη ερώτηση τώρα. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τα όρια της ΚΕΠΑ και των δράσεών τη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα των ε, ναυτικών και πώς ε, είναι συμβατό αυτό με την ρήτρα αμοιβαία συνδρομή που ορίζεται, που προδιαγράφεται στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας και ιδιαίτερα πώς συνάδει αυτό με την αντιμετώπιση των ε, προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ΚΕΠΑ. Η κυρία Λούραντσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αντίστρατηγε. Αναφερθήκατε στο CMPD και ότι έχει λάβει κάποια καθήκοντα, όπω για παράδειγμα τη διεύθυνση αντιμετώπιση κρίσεων. Υπάρχουν κάποιε ανησυχίε εδώ στο Κοινοβούλιο από διάφορε ομάδε και από το δική μου και από άλλε ομάδε όμω που απέστειλαν αποστολή, επιστολή στην Λέδη Άστον τον Ιανουάριο για το θέμα αυτό, γιατί για την υπηρεσία αυτή. Να ακούσουμε τη γνώμη σας, γιατί για παράδειγμα η μονάδα για ενοποιημένη στρατηγική, στρατηγικό σχεδιασμό που βρίσκεται υπό ε, οργάνωση. εξ όσων ξέρουμε, απαρτίζεται από άτομα με στρατιωτικό υπόβαθρο, παρά το γεγονός ότι το βασικό σκέλος είναι και στρατιωτικό και πολιτικό. Κατά 75% πιστεύετε λοιπόν ότι είναι σωστό αυτό Θεωρώ προσωπικά ότι καλύτερα θα ήταν να είχαμε μια καλύτερη διαφοροποίηση των ικανοτήτων των ατόμων του προσωπικού, γιατί όπω ξέρουμε, όλο το προσωπικό προέρχεται από το ίδιο στρατηγικό, στρατιωτικό υπόβαθρο. Αν θέλουμε λοιπόν πιο έντονο το πολιτικό σκέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια έντονη διαφοροποίηση. Και επίσης ε, για την Γενική Διεύθυνση για την Αντιμετώπιση των Κρίσεων και για την οικοδόμηση της ειρήνης εντός της υπηρεσίας αυτής. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Έλχαζον, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Μία ερώτηση. Μιλήσατε για τη στρατιωτική συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εργάζεται επί των πρωτοτύπων XUI. Το υποστηρίζετε αυτό το σχέδιο και αν ναι, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί. Ο για Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, αντιστράτηγε, να σας συγχαρώ καταρχάς για την αποστολή στην Βοσνία Ερσεγοβίνη, η οποία πραγματικά στέφτηκε με επιτυχία υπό την ηγεσία σας. Να επανέλθω στο θέμα των πειρατών, γιατί είναι ένα θέμα δημοφιλές. Δεν μιλήσατε όμως τίποτα, δεν είπατε τίποτα για τη συνεργασία με την σομαλική κυβέρνηση, με τις σομαλικές αρχέ. Υπάρχει τέτοια συνεργασία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο, κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση την γενική. Πρώτα απ' όλα μια γενική διαβεβαίωση. Με έναν ευρωσκεπτικιστή σαν και εσάς, εμείς οι ευρωενθουσια... Ευρω... προευρωπαίοι προ... πρέπει να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Μακάρι και μερικοί από εμάς να μιλούσαν από εσάς. Τώρα, ο Αντώνη Ματσάδο έλεγε σε ένα ποίημα του όποιος ξεκινάει ένα δρόμο τον διαμορφώνει ο ίδιος περπατώντας. Κάπως έτσι έγινε και η πολιτική μας. Έτσι διαμορφώθηκε. Και με την... Ε, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ και κάποια χρόνια ήταν κάτι που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί διότι υπήρχε βέτο και εκ μέρους ενός στρατηγού Άγγλου που ε, έλεγε ότι δεν ήταν ευρωπαϊκό θέμα, δεν ήταν κοινοτικό. Γι' αυτό λέγεται ότι περπατώντας κανείς διαμορφώνει την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι πραγματικότητα κυρίως με την επιχείρηση Αταλάντα. Δεν θέλω να σας κάνω καμία ερώτηση, απλώς να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε και επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Ευχαριστώ. Um, thank uh, Σας ευχαριστώ και πάλι για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Την Βοσνία Ερσεγοβίνη αν ήρθε ώρα να τερματίσουμε τις επιχειρήσεις μας. Δεν είναι στρατιωτικό θέμα. Είναι διαπίστωση στρατιωτική ότι έχουμε φέρει σε πέρας εμείς τα στρατιωτικά μας καθήκοντα, αυτά που μας είχαν ανατεθεί. Αλλά τώρα να κρίνουμε εάν θα πρέπει να είναι εκεί η στρατηγική ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα στην περιοχή είναι θέμα κρίσης των πολιτικών. Για την Κινέα Μπισάου, Γουινέα Μπισάου, εάν υπάρχει διαφορά. Η Γουινέα Μπισάου έχει τα τελευταία χρόνια τόσα προβλήματα με δολοφονίες, με δολοπλοκίες και δεν μπορώ να πω ότι εμείς κάναμε τι μεγάλη διαφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως συνεισφέραμε, διότι η κυβέρνηση και οι αξιωματούχοι ότι έχουν αρχίσει να κάνουν προτάσεις για μεταρρυθμίσεις, πράγμα που είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Και η πρόταση που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι σε ποιο ε, μέτρο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει το σχέδιο της Γουινέας Μπισάου. Αλλά νομίζω ότι όντως κάναμε τη διαφορά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια χώρα που είναι τόσο τρομερή να κάνει κάτι. Και πρέπει να πω ότι το μηδέν επί μηδέν κάνει πάντα μηδέν. Και αυτό θα μπορούσα να πω για να χαρακτηρίσω αυτή τη χώρα. Τώρα. Issue, uh, um, Για τα θέματα ναυτικών επιχειρήσεων και την, ε, τους περιορισμούς της ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Είπε η, στο τέλος των παρατηρήσεων στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα η κυρία Άστον δεν παραθέτω, αλλά είπε περίπου ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην έχουμε τεχνητά σύνορα μεταξύ του τι ακριβώς συμβαίνει εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έννοια προσπαθώ να αποδώσω. Εάν Φερρυπίν, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι είναι ένα πρόβλημα ασφαλείας, ένα ε, πρόβλημα στρατιωτικό, η κυβερνοεπίθεση είναι στρατιωτικό ή πολιτικό πρόβλημα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχει πάντα ένας ε, τομέας ε, σύγχυσης, ο οποίος όλο και περισσότερο διευρύνεται. Και στον τομέα των ναυτικών επιχειρήσεων ε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα διότι με τα ίδια μέσα πρέπει να πολεμήσουμε πολλές διαφορετικές καταστάσεις αν θέλετε. Και ελπίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε με τις ναυτικές δυνατότητες που διαθέτουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο με πολλούς τρόπους. Ίσως μπορεί να μας βοηθήσει από οργανωτικής πλευράς η συνθήκη της Λισαβόνας. Ήταν πολύ πιο δύσκολα με τους τρεις πυλώνες προηγουμένως τα πράγματα. Τώρα, η CNPD, αυτή η Γενική Διάθεση Σχεδιασμού, είναι πολύ ε, νωρίς να την κρίνουμε διότι συστάθηκε πριν από ένα μήνα, την 1η Φεβρουαρίου. Μετά από έξι εβδομάδες λοιπόν είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε κρίσεις. Η CNPD θα χρειαστεί τον υπόλοιπο χρόνο για να μπορέσει ως εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συσταθεί και να οργανωθεί. Δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε απομονωμένα, διότι θα πρέπει με συνολικό τρόπο να μπορέσει να συνεργαστεί και με όλους τους άλλους τους πρωταγωνιστές. Και θα πρέπει να δούμε όλα τα μέσα διαχείρισης κρίσεως ε, σφαιρικά σε σχέση με αυτή την υπηρεσία, σε σχέση με αυτή την διεύθυνση και την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Πολλές φορές ακόμη και στο ε, μεταξύ των στρατιωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, έχουμε επαρκή άτομα για να κάνουμε την δουλειά μας. Δεν έχουμε επαρκή και χρειάστηκε πολλές φορές να ζητήσουμε την βοήθεια για την οργάνωση και προγραμματισμό εκτός στρατιωτικών. Είναι πολύ νωρί λοιπόν να εκφράσουμε οποιοδήποτε κρίση και θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά και όχι μόνο σε ένα μέρος του τμήματος διαχείρισης κρίσεων αν χρειαζόμαστε μία ε, γενική διεύθυνση για την ε, διασφάλιση της ειρήνης. Και πάλι αυτό το θέμα θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά. Η καλύτερη κατάσταση για τους στρατιωτικούς θα ήταν να μην χρειάζεται ποτέ να μάχονται, να βρίσκονται πάντα σε κατάσταση ειρήνης. Και όταν κάνουν ειρηνευτικές αποστολές ή άλλες αποστολές ε, προληπτικά για να μην υπάρξουν συγκρούσεις, τόσο το καλύτερο. Όλα όσα γίνονται κατά την άποψή μου είναι για να μπορέσει να διασφαλιστεί και να επικρατήσει τη η ειρήνη και να μην υπάρχουν ε, εκρεμείς διαμάχες και συγκρούσεις. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενεργούμε προληπτικά για να μην φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Προσπάθησα να ακούσω και τα αγγλικά και τα γερμανικά. Το μόνο που ε, κατάλαβα ήταν η λέξη πρωτότυπο. Δεν έβαλα έγκαιρα τα ακουστικά μου. Τι ακριβώ ρωτήσατε. Μιλάμε για τα πρωτότυπα XUI, για αυτό το κοινά τυποποιημένο ε, interface χρηστών. Um, Πρόκειται. Δεν είμαι βέβαιος για ποιον τομέα αναφέρεστε. Είναι τεχνικό για μένα και δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσεις. Και τέλος, τι μορφές συνεργασίας θα έχουμε και με την κυβέρνηση της Σομαλίας